θα είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έκθεση Ουγγουρεάνου για την κινητικότητα των εργαζομένων. Τέσσερα λεπτά έχει ο εισηγητής τώρα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η μετακίνηση των εργαζομένων είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Τελικά θα διαμορφώσει το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εισηγητής θα πρέπει να κοιτάξω με θάρρο αυτή την κατάσταση που είναι ε, οικονομικά δυσβάσταχτη και μη παραδεκτή από κοινωνική απόψεω. Είναι δικαίωμα των εργαζομένων να μετακινούνται. Είναι ένα δικαίωμα που, ε, στο, με το οποίο έχουν, συμφωνήσει όλα τα κράτη-μέλη. Παρόλα αυτά, αποφασίζουν τα κράτη-μέλη να εισάγουν, να επανεισάγουν περιορισμούς ή και να προτείνουν ότι θα ανακοινώσουν και άλλα μέτρα στη συνέχεια. Αυτά ε, όλα είναι για εσωτερική πολιτική ε, κατανάλωση σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, τα οικονομικά στοιχεία είναι ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ε, στοιχεία επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδείκνεων ότι η μετακίνηση των εργαζομένων δεν έφερε αύξηση ε, της ε, ανεργίας. Δεν το τονίζω και δεν διατάραξε την αγορά εργασίας του κράτους αποδοχής. Το αντίθετο, αυτή η ροή εργαζομένων έφερε η οικονομική ανάκαμψη που κυμαίνεται στο 1% περίπου του ΑΕΠ κάποιων κρατών. Αυτή η ιδέα της περισσότερες Ευρώπης είναι στη μόδα τώρα τελευταία. Τι εννοεί κανεί, εννοούμε περισσότερη Ευρώπη αλλά για λιγότερου Ευρωπαίου. Διότι ε, έχουμε μία ενιαία αγορά για το κεφάλαιο και για τα αγαθά. Αλλά δεν έχουμε για την ε, εργασία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πως ε, οι δυτικέ επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ανατολή με επιτυχία ενίοτε ε, ε, και κάποιες φορές ε, ε, Καταργώντα χιλιάδε ε, θέσει απασχόληση, ενώ το αντίστροφο δεν μπορεί να συμβεί. Οι εργαζόμενοι από τι ανατολικές ε, χώρε δεν μπορούν να εργαστούν στι δυτικέ. Και όχι μόνο αυτό. Οι δυτικέ χώρε που παρεμποδίζουν του πολίτε των ανατολικών χωρών, συγκεκριμένα της Ρουμανία και της Βουλγαρίας, έχουν τα καλύτερα, τις καλύτερες προσφορές στην, στις ανατολικές Κατέχουν τι καλύτερε θέσει απασχόληση. Πρόκειται για μηχανικού συστημάτων πληροφορική, για δικηγόρου, για γιατρού. Ηθικώ πώ είναι εσφαλμένο αυτό και πρέπει να σταματήσει. Και ξέρετε, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα ε, να το κάνουν αυτό. Έχουν δικαίωμα να μετακινούνται και γι' αυτό υποστηρίχθηκε η έκθεσή μου. Φαίνεται αυτό από την έκθεση ψηφοφορία στην Επιτροπή και ελπίζω να υποστηριχθεί από ολόκληρο το Κοινοβούλιο στην αυριανή ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ora iniziamo il catch di AI. Catch di AI. Κυρία Ιβάνοβα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Στα αγγλικά. Θα ήθελα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 Разчитаме именно на вас да пазите и гарантирате една от основните европейски ценности. Συγγνώμη, θα πρέπει να σταματήσετε, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, μετάφραση της ομιλίας σας. Ένα λεπτάκι. Μπορείτε να ξαναρχίσετε. Εγώ ήθελα να απευθύνω έκκληση στον Επίτροπο και στην Επιτροπή να είστε αυστηροί και αντικειμενικοί όταν αναλύετε τους λόγους για τους οποίους τα διάφορα κράτη-μέλη θέλουν να υποβάλουν περιορισμούς. Πρέπει όμως πάντοτε να εγγυόμεθα τις ε, αξίες, τις ευρωπαϊκές αξίες, ελευθερία στην κινητικότητα όλων των πολιτών η κυρία Πίνκεβιτσούτε Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Ουγγουρεάνο. Η κύρια ιδέα εδώ είναι ότι η κινητικότητα των εργαζομένων είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προαχθεί. Αλλά πρέπει να προαγάγουμε μια σφαιρική ολοκληρωμένη κινητικότητα των εργαζομένων. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων στο εξωτερικό θα πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματά τους και ότι δεν θα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης αυτοί οι εργαζόμενοι. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να συνεργάζονται οι συναρμόδιες, οι αρμόδιες αρχές. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι οι πολίτες οι άνθρωποι που πάνε και εργάζονται σε άλλες χώρες πρέπει να μπορούν να διατηρούν τα επαγγελματικά προσόντα τους. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν τη διαδικασία αναγνώρισης, αμοιβαία αναγνώρισης αυτών των προσόντων από πλευράς άλλων χωρών. Και βλέπουμε ότι πολλοί καταρτισμένοι και καλά εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν κάποια κράτη-μέλη λόγω κοινωνικών συνθήκων που δεν γίνονται δεκτές από αυτούς. Και θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο να αναζητήσουν λύσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και να επιληθούν ήδη σήμερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Πρόκειται για μια καλή έκθεση που υποστηρίζουν οι πράσινοι διότι το δικαίωμα διαβίωσης ε, και εργασίας σε ένα άλλο κράτος μέλος από τις βασικές ελευθερίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έπρεπε να προστατεύσουμε αυτή την ελευθερία. Από πλευράς των πρασίνων επίσης ε, θα θέλαμε να εισαγάγουμε ε, την έννοια της ορθής και εντάξει διακίνησης των εργαζομένων. Τι εννοούμε, στη Δανία έχουμε σοβαρά προβλήματα με το κοινωνικό dumping. Υπάρχουν μισθολογικέ διαφορέ. Βλέπουμε τι διαφορέ με εργαζόμενους που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη και εργάζονται στη Δανία. Δεν μπορούμε να, διχοτο... επιτρέψουμε τη διχοτόμηση τη αγορά εργασία. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να καρπώνονται κάποιοι αυτά τα ωφέλη ε, του κοινωνικού dumping. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη ρίση των κανόνων. Χρειαζόμαστε καλύτερη ενημέρωση, μεγαλύτερη συμμετοχή και ε, κυρίως τον κατάλληλο έλεγχο, έλεγχο τόσο ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις. Σας ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Τσεσκόβα. E, Σα ευχαριστώ πρόεδρε κυρίε και κύριοι. Η Επιτροπή Γυναικ Δικαιωμάτων των Γυναικών ολοκλήρωσε την γνωμοδότησή τη για αυτήν την έκθεση και εγώ ήμουνα συντάκτρια γνωμοδότηση αυτή τη γνωμοδότηση. Η κινητικότητα είναι ένα από τα κυριότερα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πεδίο καταβάλαμε πολλές προσπάθειες για να σημειωθεί πρόοδος. Όμως εξακολουθούν και υπάρχουν κάποια προβλήματα και προσκόμματα που παρακολύουν την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με την οδηγία του 2004 είδαμε ότι η εφαρμογή αυτής, η υλοποίηση αυτής της οδηγίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους οικείους, τους συγγενείς των εργαζομένων, δεν πάει καλά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για τα δικαιώματά τους και για τα δικαιώματα των οικείων, των συγγενών τους. Θα θέλω επίσης να τονίσω κάτι άλλο. Κάνουμε λόγο εδώ για την κινητικότητα. Όταν μιλάμε λοιπόν για την κινητικότητα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οι συγγενείς και οι συμβοί, γυναίκες ή άνδρες, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια πρόσβαση σε υπηρεσίες, προσπελασιμότητα σε υπηρεσίες όπως τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγία κτλ. Γι' αυτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι η Επιτροπή Επασχόλησης δέχτηκε και έλαβε υπόψη να θέσει προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση δεν μας, μπορεί να μας αφήσει να αγνοήσουμε την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ένα τρίτο περίπου των εργαζομένων σε επισφαλή κατάσταση εργασίας, με χαμηλούς μισθούς. Έχουμε 25 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως νέους και γυναίκες που τους αρνούνται ένα μέλλον με αξιοπρεπή διαβίωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κάνουμε λόγο για κίνητρα κινητικότητας για εργαζόμενους σε πολλές περιπτώσεις σημαίνει να δίνουμε κίνητρα για το κοινωνικό dumping, την επιδίνωση της εκμετάλλευσης. Γιατί εκείνοι που σε σχέση με τις ανάγκες κάποιων που πάνε σε μια άλλη χώρα να εργαστούν εκτός της δικής τους και γι' αυτό εμένουμε και επιμένουμε σε μια πολιτική ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου ώστε στο τέλος τέλος να σταματήσουν οι πολιτικές περικοπών και λιτότητας που επιδεινώνουν τη φτώχεια και την εκμετάλλευση <clears throat> και που αφήνουν τους εργαζόμενους χωρίς καμιά δυνατότητα υπεράσπισης και άμυνας της ζωής τους και των οικογενειών τους. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε συνάδελφοι, αλλά 15 ζήτησαν το λόγο με το Catch Λοιπόν, θα περιοριστώ να δώσω το λόγο σε έναν ομιλητή. Περιορίστηκα να δώσω το λόγο σε έναν ομιλητή από κάτι πολιτική ομάδα. Ο Επίτροπος Άντορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα αρχίζοντα να ευχαριστήσω τον κύριο Τράιαν Ογκουρεάνο για την έκθεσή του σχετικά με την πρόθεση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ένωση. Σημεριζόμαστε την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με το σημαντικό αντίκτυπο που έχει η κινητικότητα επί της οικονομικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 40 χρόνια. Ε, αυτή η βασική ελευθερία διακίνησης ε, των εργαζομένων ε, ενίσχυσε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς. Επίσης, η γεωγραφική κινητικότητα τονώνει και την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία φυσικά όταν υψηλά επίπεδα ανεργίας συνυπάρχουν με μεγάλα ποσοστά φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες για να αρχίσουν ε, με αυτοπεποίθηση την σταδιοδρομία τους ε, σε ένα άλλο κράτο μέλο. Χρειάζονται καλή γνώση αγορά εργασία σε κάθε κράτος. Πρέπει να γνωρίζουν ακριβώ ποια είναι η θέση που θα καταλάβουν. Αυτό συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και δεν έχουμε περιοριστεί σε λόγια. Έχουμε εκπονήσει ε, νέα εργαλεία όπω παραδείγματο χάρη το δίκτυο παρακολούθηση των θέσεων απασχόληση. Έτσι επίσης θα ενισχυθεί και η λειτουργία του δικτύου EURES ε, που παρέχει υψηλή ποιότητα σε πληροφορίες, ενημέρωση καθώς και υπηρεσίες πρόσληψης για ε, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων του χρόνου. Ε, θα αναβαθμιστεί το δίκτυο Γιούρε για να συμπεριλάβει περισσότερες θέσεις απασχόλησης ε, όπως ανακοίνωσε εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό της σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας. Επιτροπής ε, ε, αρχίσει ε, να λειτουργεί επικυροποιημένη εκδοχή. Θα δούμε αυτά αποτελέσματα. Τώρα βρίσκεται σε πειραματική φάση αυτό το δίκτυο. Επίσης, χρειαζόμαστε καλύτερους διάβλους ε, επικοινωνίας, ε, δηλαδή ανάμεσα στις ε, κρατικές αρχές και τους εργαζομένους, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και από αυτή την πλευρά και μετά την κατάθεση της έκθεσής σας εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσθέσουμε νέες διαστάσεις στο σχέδιο σχετικά με την ισότιμη μεταχείριση των των εργαζομένων. Επίσης, θέλουμε να υλοποιηθεί καλύτερα η οδηγία του 2004 υπαριθμών 38 σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων μετά από ανησυχίες που εκφράστηκαν για αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη σημαντικά επιτεύγματα μετά από αυτές τις προσπάθειες. Πολλά κράτη-μέλη έχουν τροποποιήσει ήδη την ομοθεσία τους ή έχουν ανακοινώσει τις μεταρρυθμίσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα για να ε, εξασφαλίσουν την σωστή εφαρμογή εφαρμογή οδηγία σε περικινητικότητας των εργαζομένων. Επίση, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τι πράξει προσχώρηση ε, για τα κράτη ε, που ε, προσωρινά έχουν επιλέξει να περιορίσουν την κινητικότητα των εργαζομένων και μετά από αιτήσει τη Ρουμανία και τη σε βάσει τη πράξη προσχώρηση του 2005 πριν το τέλο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει νέα έκθεση που θα προβλέπει τι μεταβατικέ διατάξει ούτω ώστε να λειτουργήσει η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και για αυτές ε, τις χώρες. Ε, ο στόχος είναι η διαχείριση της ροής ε, των εργαζομένων για να σταθμιστεί ο αντίκτυπος που έχει στην αγορά εργασίας των κρατών μελών. Οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην τρίτη φάση, δηλαδή από την πρώτη πρώτου του 2012 και μετά κατά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι θέμα των κρατών μελών. Θα πρέπει να καταβάλουν τι απαιτούμενε κοινοποιήσει ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, σημειώνονται σοβαρέ διαταράξει ε, στην αγορά εργασία. Του. Καλωσορίζουμε την έκθεση πρωτοβουλία που υποβάλλατε και επιβεβαιώνουμε και πάλι ότι πρόκειται εδώ για μια πρωταρχική ελευθερία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είναι αδύρυτη ανάγκη να προωθήσουμε την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων διότι αυτό θα τονώσει και τι οικονομίε μα κυρίω τώρα που παρατηρείται θεωρείται εντελώ ετεροβαρή σε οικονομική ανάπτυξη. Εξάλλου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020 που έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ Επίτροπε. Πέρα στη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30.